die Präsidentin. Einen schönen guten Nacht. Καλό σας απόγευμα. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, πριν ε, μπω στα σημεία τη της θα ήθελα να ε, ενημερώσω για όσους δεν το άκουσαν ότι σήμερα και πάλι να βάγισε νοτίως της Σικελίας ένα ε, πλοίο γεμάτο πρόσφυγες που μάλλον είναι και εκατοντάδες τα θύματα που θρυνούμε. Και θα ήθελα να πω ότι εμείς ως Κοινοβούλιο διαπιστώνουμε ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, επαναλαμβάνονται το τελευταίο διάστημα, μήνες τώρα. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις και θα φροντίσουμε τέτοιου είδους δράματα να μην ξανασυμβούν γύρω από την Ήπειρό μας. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στα πρακτικά, τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινή συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, δεν έχετε... Ε, εγκρίνονται τα συνοπτικά πρακτικά. Έχω μια ανακοίνωση να σας κάνω από